Υπάρχουν ανακοινώσεις. Στα τσεχικά θα τις κάνω. Η Επιτροπή η Νομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού, έχει δώσει εντολή στον κύριο Ζόλταν Μπαγκόα, για να έρθει στις 12 Σεπτεμβρίου του 10 να εγκριθεί μάλλον ο ορισμός του. Είναι κανείς κατά, όχι εγκρίνονται τα διαπιστευτήριά του. Τα πρακτικά της συνεδρινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου. Και τότε θα εγκριθούν και θα σταλούν στους δικαιούχους. Λίγοι εδώ προσωρινά διακόπτεται η σύνοδος και σας εύχομαι καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε.